Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, πέραν της ε, περιπτώσεις του Φαραή Βαγκού υπάρχει η περίπτωση της εκμεταλλεύσεως των διαμαντιών υπάρχει η διαδικασία του Κίμπερλε και ε, επιτρέπονται να πολλούνται τα διαμάντια αρκεί να μην χρηματοδοτούν τις ένοπλες σειράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία του Κίμπερλι στην τελευταία συνάντηση 21 με 23 Ιουνίου δεν μπόρεσαν οι συμμετέχοντες να ε, καταλήξουν σε συνένεση για την πιθανή προσθήκη των δυσμάτων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στη ε, δικασία του Κίμπερλι και υπάρχουν παραβιάσεις από τις υπηρεσίες πληροφοριών εκ των οποίων ε, ένας ε, υπεύθυνος ήταν ο Φαράι Μαγκού, ο πολίτης της Ζιμπάμπουε και ιδρυτής διευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης και συνελήφθη στη Ζιμπάμπουε διότι λέγεται ότι είχε παραβιάσει την ασφάλεια του κράτους Ζητούμε λοιπόν να αποστρατικοποιηθεί η εκμετάλλευση διαμαντιών, να ε, ισχύσει η διαδικασία του Κίμπερλε και να μοιραστεί τους λαούς ο πλούτος του Κίμπερλε μέσω ε, ενός ε, κυριάρχου ταμείου για να μπορέσουν να ισχύσουν τα δικαιώματα δημοκρατίας και ελευθερίας στις χώρες αυτές και να ενισχύσουν με την ε, συζήτηση που έχουμε με το Ζιμπάμπουε. Η κυρία Τζοντίνη για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, δύο πράγματα διακυβεύονται. Πρώτα απ' όλα το πρόβλημα αυτό καθεαυτό και το άτομο. Το άτομο Φαράι Μαγιού ήταν ε, ε, υπέρμαχος των δικαιωμάτων που συνελήφθη στο Ζιμπάμπου και μετά τον κακομεταχειρίστηκαν στη φυλακή. το παρατηρητήριο της διαδικασίας του Κίμπερλεϊ που πρέπει να παρακολουθεί την κατάσταση στο, στο Ζιμπάμπουε παίζει παράξενο ρόλο. Ήρθε σε επαφή με τις αρχές του Ζιμπάμπουε και χρησιμοποίησε τις πληροφορίες που παρέλαβε από τον κύριο Μαγκού και αυτό περιέπλεξε ακόμα περισσότερο την κατάσταση του κυρίου αυτού. Και μετά είναι και ποιο είναι ο ρόλος της διαδικασίας του Κίμπερλι. Εγώ ήμουν μέλο λόμπι για μια οργάνωση ανάπτυξη που συμμετείχε στι διαδικασίε. και δημιούργησε και αυτή αυτό το σύστημα. Το σύστημα λειτουργεί, επέτρεψε πόλεμοι στο Κογκό, στην Αγκόλα, στη Σιέρα Λεόνε, να χρηματοδοτούνται λιγότερο από τα χρήματα των διαμαντιών. Τώρα διατρέχουμε τον κίνδυνο όλο το σύστημα Κίμπερλι να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς, δηλαδή για την ε, εκμετάλλευση των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη δίωξή τους. Και αυτό ζητάμε να αλλάξει το σύστημα. Από το ψήφισμά μας, το ψήφισμά μας λέμε ότι τα διαμάντια του αίματος της σύγκρουσης είναι κάτι ε, διαφορετικό από απλές πέτρες πολύτιμους λίθους. Είναι λίθοι οι οποίοι ε, γίνονται δικείμενο εκμετάλλευση σκοπού που δεν μπορούμε να δεχτούμε. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τη Ζιμπάμπουε αλλά και για την Αγγόλα και για άλλε χώρε. Γιατί δεν λειτουργούν τα πράγματα τώρα. Το σύστημα του Κίμπερλεϊ είναι ένα σύστημα το οποίο συναθρίζει πολλές χώρες ε, και δεν κινείται πολύ ομοιόβορθα. Θα πρέπει να αλλάξουμε την κατάσταση μέσα του ψηφίσματό μας. Κύριε ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι επιτέλους κάποια ησυχία και ηρεμία εδώ σε σχέση με αυτά που γίνανε το πρωί. Ε, επέβαλα το ψήφισμα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ζιμπάμπουε και το περίπτωση Φαράη Μογκαμπού, διότι δεν μπορεί να σιωπά το Κοινοβούλιο ένα τη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών που διαπράττονται εδώ και πολλέ δεκαετίε στη Ζιμπάμπουε. Ο διευθυντή του Κέντρου Έρευνα και Ανάπτυξη, ο Φαράη Μουγκάμπου, συνελήφθη από τις αρχές της χώρας του που κατήγγειλε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στα δαμαντορυχεία απλώς άσκησε το δικαίωμα της, της ελευθερίας του λόγου και το δικαίωμά του να ζητήσει πληροφορίες τα δικαιώματα το, τα ανθρώπινα και όλες τα ελευθερίας. Ζητά την απελευθέρωσή του Κοινοβούλιο και το σεβασμό της Ζιμπάμπου των πολιτικών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, ώστε να επιτρεπεί στην κοινωνία των πολιτών να εκφράζεται χωρίς φόβο. Το Ζιμπάμπουε θα πρέπει να σέβεται τι δεσμεύσει που έχει αναλάβει στα διαδικασία του Κίμπερλι και λεπτομερώ όσον αφορά την παραγωγή διαμαντιών, ούτω ώστε να βγούμε από τον φαύλο κύκλο αυτό τη χρηματοδοτήσεω ενόπλων σειράξεων. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Βερζιάτ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βλέπω ότι το ημικύκλιο είναι ήρεμο, αλλά λυπούμε που δεν είμαστε περισσότεροι που να ενδιαφερόμαστε για αυτά τα θέματα, διότι η κατάσταση στη Ζιμπάμπου είναι δραματική και αυτό δεν το εκφράζει επαρκώς το τι συμβαίνει διότι ε, δεν υπάρχει δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Οι τελευταίες εκλογές έγιναν σε κλίμα τρομοκρατίας και ε, μετά από μία συζήτηση με τον κύριο Σίκαν, τον ε, επόπτη του Κίμπερλε, είναι απλώς ένα επιπλέον επεισόδιο στη μακριά λίστα παραβιάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, υπάρχουν ε, τραγικές συνθήκες στα δαμαντορυχεία ε, δολοφονίες, βασανιστήρια ε, προς όφελος των φίλων του κυρίου Μουγκάμπε. Πολλές φορές οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις το έχουν καταγγείλει και μεταξύ αυτών η οργάνωση του κυρίου Μαγκούβου οπότε είναι περίεργο ότι ο κύριος Σικάνα αναφέρεται εις την ε, συμμόρφωση της χώρας στη διαδικασία του Κίμπελε διότι ε, δεν μπόρεσε η διάσκεψη του Τελαβίβ να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, λήψη συνενέσεως δεν πρέπει να, ε, ε, να ξαναξεκινήσει τις εισαγωγές διαμαντιών από τη Ζιμπάμπουε και θα συνεχίσει να μάχεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσει το κράτος να εμποδίσει την εισαγωγή διαμαντιών από το Ζιμπάμπουε όσο υπάρχει κράτος τρομοκρατίας. Ε, μπορεί... Γιατί στηρίξατε τον κύριο Σικάν να δώσει το πράσινο φως εφόσον ένα μέρος των σημειώσεών του είχαν ε, ληφθεί από ε, τα, τις αποσκευές του στο Ζιμπάμπουε. Πρέπει να υπάρχει μία σταθερή θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θα παρακαλούσα να μας πείτε ποια θα είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο, στην Αγία Πετρούπολη. Ο κύριος Βανόρντεν για 1,5 λεπτό. Από όταν εξελέγει το 1999 έκανα το περισσότερο για να ε, να αντιταχθεί στην αδικία το κοινοβούλιο κατά του Μουγκάμπουε και κατά των διαφόρων υποστηρικτών του που εστάφη κατά του λαού του Ζιμπάμπουε. Εδώ το κοινοβούλιο μιλά ενωμένο. Εδώ μιλάμε για συστηματική κατάχρηση των εργαζομένων στα δαματορυχεία τη Ζιμπάμπουε από τι δυνάμει ασφαλεία του κράτου. Το Ζιμπάμπουε είναι πλήρε μέλο τη διαδικασία του Κίμπερλι, τον άτυπο φορέα που, διεθε... που ρυθμίζει το παγκόσμιο εμπόριο σε κατέργα διαμάντια. Και μέχρι τώρα δεν έκανε πολλά πράγματα για να σταματήσει τι καταχρήσει. Καλό τη διαδικασία τη Κίμπερλι να λάβει σκληρά μέτρα κατά τη Ζιμπάμπουε, διότι δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα αυτά τη συμφωνία. Καταδικάζω και εγώ τη σύλληψη του κ. Μαγκούβου, ο οποίο. Είναι άνθρωπος με συνείδηση και κατήγγειλε τις βίαιες πράξεις των δυνάμεων ασφαλείας ε, ε, του Ζιμπάμπου. Η κυβέρνηση της Ζιμπάμπου θα πρέπει να απελευθερώσει αμέσως τον κύριο Μαγκούβου και όλους τους άλλους πολιτικούς κρατωμένους και θα πρέπει αυτό να το επενθυμίσουμε. Το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου ήταν μια από τις βασικές δεσμεύσεις που ανέλαβαν όλα τα μέρη στην παγκόσμια αυτή συμφωνία πέρσι. Για την ώρα, οι ιατρικές ανάγκες και οι βασικές ανάγκες μεγάλου τμήματος του πληθυσμού της Ζιμπάμπουε καλύπτεται από διεθνή βοήθεια. Η κυβέρνηση Ζιμπάμπουε θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το σημαντικό εισόδημα από τα δαμαντορυχεία για να δημιουργήσει ένα ταμείο για τα δαμάτια. για να προωθηθεί η οικονομία και να παραχθεί κοινωνική χρηματοδότηση, παιδεία και υγεία να καλύπτεται αυτά που καλύπτονται τώρα από του διεθνεί δωρητέ. Δυστυχώ, κυρία Πρόεδρε, έχει πολύ δρόμο το Ζιμπάμπε μέχρι να πούμε ότι ο λαό τη ζει ελεύθερα και δημοκρατικά ε, και σε πλαίσια κράτου δικαίου. Είναι η ώρα για δραματικέ αλλαγέ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρε τη Νοτιού Αφρική θα πρέπει να πιέσουν περισσότερο την κυβέρνηση, ώστε να υπάρχει ορθή διακυβέρνηση στη Ζιμπάμπουε. Και τώρα ο κ. Γκάλερ, για ένα λεπτό, είναι εξάρτητοι αγορητέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τον κύριο Μαγκούβου και τις δημοσιεύσεις του που οδήγησαν εις τη σύλληψή του για την εκμετάλλευση της περιοχής του Μαράγκε δείχνει ε, ποιος έχει την εξουσία αυτή την εποχή στο Ζιμπάμπουε και ότι η κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητος ε, είναι μια καταναγκαστική ε, κυβέρνηση συνασπισμού ε, και απλώς ο Μουγκάμπε εξασκεί μέσω αυτής την εξουσία του και γι' αυτό συνεχίζονται αυτές οι καταστάσεις και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ε, εφαρμόσουμε ε, τον κατάλογο ε, που έχουμε αυτών που δεν ακολουθούν τις αρχές μας θα έπρεπε να πούμε ότι τα αποτελέσματα της πωλήσεως των διαμαντιών διατίθενται σε λίγους και όχι σε όλους, όλους τους πολίτες της χώρας που τα δημιουργούν. Οπότε ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νότιος Αφρική πρέπει να κινηθούν για να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Ο κύριος Κάσμαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βελτιώθηκαν τα πράγματα στο Ζιμπουάμπο, αλλά δυστυχώς δεν βελτιώθηκαν αρκετά την καταπίεση του κ. Μαγκούβου και των άλλων υπερασπιστών των δικαιωμάτων και είδαμε ότι έκλεισαν και συνέλαβαν τους αμφιφιλόφιλους ε, και ομοφιλόφιλους ε, στη χώρα. Λοιπόν, τώρα που μιλώ ως Άγγλος, θα το απέριπταν αυτό που λέω. Σαν Ευρωπαίοι θα απέριπταν εμάς αυτά που λέμε. Τι είναι προφανές για τις αφρικανικές χώρες, τι έχω να τους πω. Ξέρετε τι συμβαίνει στη Ζιμπάμπουε. Και αυτό που συμβαίνει είναι λάθος. Αν δεν κάνετε κάτι μαζί, θα χάσετε η αδίποτε ηθική πυγμή στην Ήπειρο και στον κόσμο. Η Αφρική είναι στα χέρια σας. Το μέλλον της Αφρικής στα χέρια σας. Το να κάθεστε με σταυρωμένα τα χέρια ενώ συλλαμβάνεται κόσμο, διότι θέλει να εκθέσει παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να υπερασπιστεί τι απλέ γυναίκε και του άντρε, εάν δεν κάνετε τίποτα, Αφρική θα είναι σαν να είσαστε συνένοχοι. Ευχαριστώ κύριο Σκάλ, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Προσπαθούμε πάντα να είμαστε αποτελεσματικοί και να παρεμβαίνουμε όσον αφορά τα θέματα αυτά σαν Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπο έξυπνο να πιέσουμε το καθεστώς Μουγκάμπε. ούτως ώστε να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα όπως συνέβησαν στον κύριο Μαγκούβο. Το θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κάτι που αφορά την θεμελιώδη αξιοπιστία της χώρας. Θα πρέπει να λέμε αν τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται σεβαστά ή όχι. Δεν θα πρέπει να αρκούμαστε και να ικανοποιούμε θα μικρές πρόοδους. Δεν πρέπει να αρκούμαστε στα λίγα. Πρέπει να λέμε σαφώς ότι η κυβέρνηση του Μουγκάμπε δεν έχει νομιμότητα. Και θα πρέπει αυτό να το πούμε ξάστερα, ξεκάθαρα. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Πρέντα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ζητήσω την άμεση απελευθέρωση του Φαρουάη Μουγκάμπε και θα ήθελα τα δικαιώματά του να γίνονται σεβαστά. Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών είναι πολύ σημαντικός, όχι μόνο η διαδικασία Κίμπερλεϊ, αλλά και για την ε, παγίωση της δημοκρατίας στη Ζιμπάμπουε. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι γίνεται πρόοδο, σημειώνεται πρόοδο όταν οι υπασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φημώνονται, όταν προσπαθούν να ειδοποιήσουν τα διεθνή μέσα ενημέρωση για παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να υπογραμμίσω επίσης ότι οι αρχές της Ζιμπάμπουε πρέπει με αμερόληπτο τρόπο να αντιμετωπίζουν τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων αυτών που σημειώνται στα δαματορυχεία. Βασική λέξη, λέξη κλειδί είναι η διαφάνεια. Οι πολίτες της Ζιμπάμπουε έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται και οι αρχές θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις δεσμεύσεις που εφεδροντικά ανέλαβαν. Ευχαριστώ Γκόμες για ένα λεπτό. Κυρία Γκόμες. Η υπόθεση Φαράγε Μαγκούβου δείχνει ποια είναι η κατάσταση στη Ζιμπάμπε και ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η διαδικασία του Κίμπερλι. Δεν θα χρησιμοποιούνται τα διαμάντια ε, για πόλεμο, θα πρέπει να καθαριστούν παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από τη χρήση του για τον πόλεμο. Θα και αυτό εξαρτάται και επίση και από τι εταιρείε που εκμεταλλεύονται τα θεματορχεία. Τα διαμάντια είναι σημαντικά για να καταπολεθεί η φτώχεια και να επιτευχθούν οι στόχοι τη χιλιετία. 293 δισεκατομμύρια δολάρια πετρελαίου εξήγαγε η Αφρική το 2008 ε, που είναι μεγάλο ποσοστό της βοήθειας που δέχεται, πολύ μεγαλύτερο. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε το κράτος δικαίου, την ε, κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων για να υπάρχει ε, ευμάρεια στην Αφρική και το σεβασμό των θεμελιών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να δώσει του κατάλληλου μηχανισμού Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση αυθορά στα ανθρακοριχεία. Όπω είπαν πολλοί βουλευτέ, Υπάρχει το www.stopcorruption.eu ε, και υπάρχει εκεί μια αίτηση που παρακαλούμε να την υπογράψετε. Ευχαριστώ και πάμε στον κύριο Ομπερμάιερ. Μην γεγραμμένος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι πολύ ευτυχής ότι μιλάμε σήμερα για την περίπτωση Μαγκούβου που είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου διότι ο Μουγκάμπε ήταν ε, κάποτε ένας υπερασπιστής των δικαιωμάτων των μαύρων και τώρα είναι ένας στιγνός δικτάτορας ε, στην τελευταία εποχή διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό των ανέργων στη χώρα αυτή είναι τεράστιο. Ποιος φυλακίζει και βασανίζει και ε, απειλεί τις οικογένειες ε, ποιος δεν σέβεται ε, την ε, διαδικασία του Κίμπελη αλλά σύμφωνα με τη διαδικασία του Κίμπελη πρέπει να προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και αντί να γκρινιάζουμε εδώ και να παραπονιόμαστε θα έπρεπε να επιβάλλουμε κυρώσεις στη Ζιμπάμπουε για να μπορέσει να συμμορφωθεί στη διαδικασία του Κίμπελη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επανέρχομαι τώρα στους μεμονωμένους ομιλητές, τον κύριο Κασμάρεκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρουμε όλοι ότι τα διαμάντια μπορούν να είναι και ευλογία και ε, μάστιγα και θα θέλαμε να υπάρξει μια αλλαγή των δομών στη χώρα αυτή κατά τρόπον ώστε να υπάρξει μια θετική εξέλιξη. Σήμερα μιλάμε για κάποιον για τον οποίο τα διαμάντια ε, μπορεί να αποδειχθούν σαν ε, ένα αρνηστικό στοιχείο διότι ε, σαν αρχηγός μια μιας, ανθρώπινης, μιας οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει διαπιστώσει πολλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βλέπουμε ότι αυτοί οι οποίοι πληρώνται σπεσμένα δεν είναι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται. Ελπίζω λοιπόν ότι κάποια στιγμή η κυβέρνηση της χώρας αυτή θα ακούσει τη φωνή μας διότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δαμαντορυχεία αυτά για μια θετική εξέλιξη ανάπτυξη της χώρας και θα ήταν καλύτερα τα κέρδη από τα διαμάντια να χρησιμοποιηθούν για την υγεία και την προώθηση της χώρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Η περίπτωση που συζητάμε εδώ σήμερα, δηλαδή η σύλληψη του κυρίου Μαγκούβου, δείχνει ότι δεν υπάρχει πρόοδος στη Ζιμπάμπη όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ελκύει την προσοχή στη σοβαρότατη κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των δεδομοντορχείων όπου κατηγορείται ο στρατός για παραβιάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Ζιμπάμπουε μπορεί να είναι σε μια κατάσταση οικονομική χρεοκοπία και τα διαμάντια του αίματο είναι απόδειξη του κινησμού των αρχών και της έλλειψης σεβασμού προς τους πολίτες τους. Το Ζιμπάμπουε παραβιάζει τους κανόνες που θεσπίστηκαν τη διαδικασία του Κιμπερλέ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθήκον να υποστηρίξει αυτή τη δομή, αυτό το σχήμα, τη διαδικασία αυτή, ούτως ώστε να καταργηθεί η κυκλοφορία και πώληση αυτών των διαμαντιών τη συγκρούσεω, των συγκρούσεων που χρηματοδοτούνται για την χρηματοδότηση συγκρούσεων. Θέλουμε ο Φαράχη Μαργκούβου να απελευθερωθεί αμέσως και απευθύνουμε έκκληση προ την ευρωπαϊκή διπλωματία, ούτω ώστε να θετήσει και να, να μάλλον αναλύσει κατά πόσο ήρθε η ώρα τώρα να υιοθετηθούν κυρώσεις κατά τη Ζιμπάμπουε και να τεθεί τέρμα στην αιματηρή αυτή κατάσταση επικρατική. Το τμήμα αυτό τη προσεκτική προσοχή του Προέδρου έχει λήξει. Μάλλον σε αυτή τη διαδικασία έχουν περισσότερου αγορητέ από ό,τι θα μπορούσαν να μιλήσουν στο ΚΑΣΤΙΑ. Ο κ. Κάλαν πρώτο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, λιγότερο από τρει εβδομάδε πέρασαν από, από τα συνελήφθηκε Μαγκούβου από τι αρχέ τη Ζιμπάμπουε και έκτοτε εκρατήθη, κρατείται μάλλον, και είναι άγνωστε συνθήκε υπό τι οποίε κρατείται και στερείται των προσωπικών, των ατομικών των δικαιωμάτων. Χαίρομαι που το κοινοβούλιο αυτό είναι ενωμένο ζητώντα την άμεση απελευθέρωση αυτού. Αλλά ανησυχώ ε, διότι η σύλληψή του ίσως να είναι ένα βήμα επαναχώρησης σε σχέση με τα αποτελέσματα της διαδικασίας του Κίμπερλεϊ. Όπως ανέφερε ο συνάδελφος Βανόρντεν, η συστηματική κατάχρηση των εργατών στα δανταματορυχεία και η κατάσταση στη Ζιμπάμπουε Μα δείχνει ποια είναι η κατάσταση στη Ζιμπάμπουε. Ότι τα τεράστια έσοδα από τα ορυκτά δεν μοιράζονται στον πληθυσμό που παραμένει φτωχό και υποφέρει από ασθένειε. Συμφωνώ επίση ότι οι αφρικανικές χώρες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση εκεί. Και υποστηρίζω το διάλογο με τη Ζιμπάμπουε από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπό τον όρο ότι ο κύριος Μουγκάβου θα απελευθερωθεί και η διαδικασία του Κίμπερλι θα πρέπει να γίνει σεβαστή από τις αρχές της Ζιμπάμπουε. Ο κύριος Τάνοκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στα 30 χρόνια από όταν ανέλαβε την εξουσία ο ο, ο κ. Μουγκάμπε έχει τελικά φτωχύνει η χώρα. Το Ζιμπάμπου τελευταία 10 χρόνια συστηματικά φτωχαίνει. οι περισσότεροι από τα 10 εκατομμύρια είναι φτωχή. Και οι φυλάρχοι του Ζιμπάμπου πλουταίνουν. Διότι εκμεταλλεύονται γέες που αρπάζουν και ορυκτά. Ε, είπε ο Μαγκάουβου που συνελήφθη ότι σκοτώνονται πάρα πολύ από το στρατό, εξώδικα και τελικά ε, τροφοδοτούνται οι φύλαρχοι του Μουγκάμπου από τα χρήματα των διαμαντιών. Άρα δεν θα πρέπει να στη δικαστική πέλη ο Μουγκάμπου, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει αυστηρέ κυρώσει εναντίον εκείνων στη Ζιμπάμπου που πλούτησαν μέσω του εμπορίου όσον αφορά τα διαμάντια αυτά του αίματο, όπω ο Καλούντου και ο Φαράχμου Μαγκούβου, που ασκούσε το θεμελιώδε δικαίωμά του τη ελευθερία του λόγου, θα πρέπει να απελευθερωθεί αμέσω από το κατετήριο. Η κυρία Κιντολεύσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε στην απόφαση του 2000 οι ε, τότε κυβερνήσεις ορισμένων χωρών είχαν κυρώσει τη διαδικασία του Κίμπελι η οποία προερχόταν από την σκέψη να σταματήσει το εμπόριο των ματωμένων διαμαντιών. Πρόκειτο από οργανώσεις ε, οι οποίες έπρεπε να σταματήσουν διότι χρηματοδοτώντουσαν ε, από την παράνομη πώληση των ε, διαμαντιών. Αλλά όλα αυτά συμβάλλουν σε προβλήματα στην Αφρική και γι' αυτό είναι ανησυχητικό ότι ε, μετά από την κατάληψη του αδαμαντορυχίου στο Μαράγκε ε, υπάρχει αυτή η κατάσταση διότι η κυβέρνηση ε, λέγει ότι προσπαθεί να αποκαταστήσει την κατάσταση και καταδικάζουμε και την σύλληψη του κυρίου Μαγούβε. Κυρίες και κύριοι, η διαδικασία του Κίμπελ είναι μια διαδικασία από εκπροσώπους των κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών για να μπορέσουν να δώσουν τέλος στα ματωμένα διαμάντια και στο εμπόριό τους αλλά βλέπουμε ότι έχει διαπιστωθεί παράνομη πώληση των προϊόντων αυτών στο Μαράγκε ε, στο Ζιμπάμπουε και ο κύριος Μαγκάουι το έχει ε, καταγγείλει οπότε βλέπουμε ότι πρέπει να ζητήσουμε να λάβει το Ζιμπάμπουε ε, τα μέσα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε, αλλά εδώ θα σταματήσει το Catch the Eye. Ήδη πήραμε περισσότερους από όσους θα έπρεπε και τώρα ζητώ από την ε, ε, Επίτροπο να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Είμαι πολύ ευχαριστημένη που διεξάγεται αυτή η συζήτηση εδώ σε αυτή την αίθουσα σήμερα. Η σύσκεψη της διαδικασίας Κίμπελη στο Τελαβίβ που έγινε στις 21 24 Ιουνίου φέτος ήταν πράγματι σκοτεινιάστηκε από τη σύλληψη του κυρίου Φαράχη Μαγκούβη, Μαγκούβου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται στι ανησυχίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επέμεινε ο κύριος Μαγκούβου να αντιμετωπιστεί νόμιμα, να μπορεί να απολαύσει τα νομιμά του δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ στην κατάστασή του, είναι σε επαφή με τους δικηγόρους του κυρίου Μαγκούβου και σκεφτόμαστε ποια στατική θα χρησιμοποιήσουμε την, ε, για να υποστηρίξουμε του ασφιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί και να βελτιώσουμε την ασφάλειά τους. Ζητήσαμε από το Ζιμπάμπου να επιβεβαιώσει το ρόλο που διαδραματίζει, ε, να ενισχύσει το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στη δικασία του Κίμπερλεϊ. Εντολή τη διαδικασία του Κίμπερλεϊ είναι να αποφευθεί το εμπόριο, να σταματήσει το εμπόριο των διαμαντίων του αίματο. Αλλά είναι σαφέ ότι αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να λειτουργήσει εν κενό αμελώντα τι ανησυχίε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό είναι ένα ισχυρότατο μήνυμα που σήμερα απεστάλλει από αυτή την αίθουσα. Έτσι δε περαιτέρω όταν αναγνωρίζουμε ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μια αρχή που βασίζει και υποστηρίζει το βασικό στόχο της διαδικασίας του Κίμπερλι. Τώρα στρεφόμενοι στη συνάντηση στο Τελαβίβ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε τη συνεχή εφαρμογή της αποφάσης του Άκαμπουντ και της ε, ούτως ώστε οι εταιρείες στο Μαράγκουε να συμμορφωθούν με τους κανόνες της διαδικασίας του Κίμπερλεϊ και την εφαρμογή του μηχανισμού εποπτευόμενων εξαγωγών. Πιστεύουμε ότι περαιτέρω συνομιλίες με το Ζιμπάμπουε στα πλαίσια διαδικασίας του Κίμπερλεϊ ε, προσφέρει την καλύτερη δυνατή λύση, όχι μόνο τόσο ώστε να εξασφαλίσουμε την τεχνική συμμόρφωση στον τομέα των ορυχείων Μαράγκε, να συμμορφωθούν με τη διαδικασία του Κίμπερλι, αλλά και να βελτιωθούν και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μαράγκε. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε τη Ζιμπάμπουε να τηρήσει τι δεσμεύσει που ανέλαβε στα πέστη δικασία του Κίμπερλι και στα πλαίσια του κοινού προγράμματο εργασία του, τόσο τα διαμάντια του Μαράγκε να μπορούν σε κάποια φάση, ανευθέτω ευθέτω χρόνο, να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη τη Ζιμπάμπουε. Στόχο μα, οι συμμετέχοντε στη δικασία του Κίμπερλεϊ και η Ζιμπάμπουε να εντατικοποιήσουν τι προσπάθειέ του, ούτω ώστε να πετύχουν συνένεση επί του δυσκόλου αυτού θέματο στο πνεύμα διαλόγου και συνεργασία. Ένα πνεύμα που πάντα διέπνεε την όλη διαδικασία. Τέλος, είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να ενημερώνεται και πρέπει να πούμε ότι συνάντηση υπουργών με υπουργού που, ε, της Ζιμπάμπουες της 2 Ιουλίου που αντιπρόσωπαν την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας η Βαρόνη Άστον, αντιπρόσωπο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είπατε εκπρόσωπος υπενθύμησε ότι η εφαρμογή της Γενικής Συμφωνίας αυτής που καλύπτει τις ανησυχίες μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, τις δημοκρατικές αρχέ είναι κλειδί για την εξομάλυνση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είπαμε στου υπουργού. Όπω είπα και προηγουμένω, προσδίδω μεγάλη σημασία στη συμμόρφωση τη Ζιμπάμπουε με του κανόνε περί κράτου δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό επανειλημμένα το έχουμε πει και σε διάφορα βήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματο... θα εξακολουθεί να χρηματοδοτεί σειρά δραστηριοτήτων εις Ζιμπάμπουε σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών, θα εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε τρόπου για να δημιουργούμε και να υποστηρίζουμε ένα ανοιχτό πολιτικό περιβάλλον. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίε γίνονται πλήρω σεβαστά. Όσον αφορά τη θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το εμπόριο ε, των διαμαντιών από τη Ζιμπάμπουε, ζητήσαμε έλεγχο των αποθεμάτων διαμαντιών πριν προχωρήσουν εσδήποτε συζητήσει για περιορισμένη επανάληψη των εξαγωγών. Καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση στην συμμετοχή των εμπλεκομένων που κάλεσε ο πρόεδρος της διαδικασίας του Κίμπερλι στα περιθώρια του Συμβουλίου για τα Διαμάντια στις, τον Ιούλιο 14 στην Αγία Πετρούπολη όπου εκεί θα προχωρήσουν περαιτέρω οι συζητήσεις όσον αφορά αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν 7 ε, ε, προτάσεις ψηφισμάτων που θα ψηφιστούν μετά τη συζήτηση. Και τώρα γυρίζουμε στο επόμενο θέμα.